Εσείς οι τίτλοι των ε, νομοθετημάτων αυτών θα δημοσιευτούν στα πρακτικά της συνεδρίασης διάσκεψη των Προέδρων σύμφωνα με το ε, άρθρο 140 του κανονισμού ε, ενέκρινε και ψήφινα το οποίο σας ε, υποβάλαμε και σας αποστήλαμε και η Ηνωμένη Αριστερά, η ομάδα της Ηνωμένης Αριστεράς κατέθεσε ένα αίτημα για την Τετάρτη αλλά για τη Δευτέρα καταρχάς, για την Δευτέρα σήμερα υπάρχουν επιθυμίες για κάποια αλλαγή της ημέρης σύνταξης, όχι για την Τρίτη παρακαλώ Δεν υπάρχει σχόλιο. Για την Τετάρτη λοιπόν η Κούε ζητήσε να συζητηθεί το θέμα της προφορικής ε, ερώτησης για το θέμα της απόφασης της Ιαπωνίας να ξαναξεκινήσει την φαλανοθυρία την περίοδο 2015-2016 και ζήτησε να υπάρξει ψήφισμα το οποίο και θα ψηφιστεί κατά τη διάρκεια της Συνόδου του Ιουλίου. Η κυρία Χάζεκαμ θα πάρει το λόγο να αιτιολογήσει το αίτημα αυτό. Παρακαλώ έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να σας ζητήσω να προσθέσουμε ένα ψήφισμα μετά την προφορική ερώτηση για την φαλανθυρία της Ιαπωνίας και να ψηφίσουμε το ψήφισμα αυτό στην Ολομέλεια του Ιουλίου. Η Ιαπωνία τους τα επόμενα χρόνια θέλει να πιάσει, να σκοτώσει, να φυλακίσει, όπως θέλετε, παιδί του, 4.000 φάλαινες από τον Ειρηνικό ωκεανό. Απειλούνται από την ε, αλληλεία της Ιαπωνία πάρα πολλά είδη. Πρόκειται για το δεύτερο μεγαλύτερο ζώο ε, του πλανήτη μας, η φάλαινα, το οποίο απειλείται με εξαφάνιση και ισχύει η σύμφωνη του 1980 για την απαγόρευση της φαλανθερία, αλλά αγνοεί επιτεκτικά η Ιαπωνία και άλλες χώρες αυτή την σύμβαση. κοιτώντα λοιπόν πώς εξαφανίζονται οι τελευταίες φάλανες, αυτό θα κάνουμε από πλευρά του Κοινοβουλίου ή θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μα για να το αποτρέψουμε. Εγώ το τελευταίο επιλέγω. Ελπίζω και εσεί το ίδιο. Θα ήθελε, λέει ο Πρόεδρο, ε, σα ευχαριστούμε. Θα ήθελε κάποιο να πάρει το λόγο υπέρ του αιτήματο που εξέφρασε η κυρία Χάζενκαμ, ο συνάδελφο Λάμπερτ. Κύριε Πρόεδρε, αύριο θα συζητήσουμε στην ομάδα για το θέμα αυτό και μιλάμε για τις φάλαινες, το μεγαλύτερο θηλαστικό που βρίσκεται ακόμη εν ζωή στον πλανήτη μας, ενώ τόσα είδη χάνονται το ένα μετά το άλλο. Είναι σημαντικό λοιπόν ε, το κοινοβούλιο μας να συζητήσει αυτό το τόσο σημαντικό θέμα για την βιοπικιλότητα. Ευχαριστώ. Θα ήθελε κανείς να πάρει το λόγο κατά του αιτήματο αυτού. Κανείς. Ας ψηφίσουμε. Με ονομαστική κλίση όπως και ζητήθηκε. Ποιος είναι λοιπόν υπέρ του αιτήματο τη κυρία Χάζε Κάμπο. Χαιρόμαστε και κλείσει, διορθώνει ο πρόεδρο. Έναρξη ψηφοφορία. Εάν ψηφίσατε όλοι. Άλλη μια φορά ρωτώ. Ψηφίσατε παρακαλώ όλοι. Πέρας. Πέρας ψηφοφορίας. Το αίτημα εγκρίνεται. E για την Πέμπτη το ΕΛΚ ζήτησε ε, να μετακινηθεί από το πρωί στο απόγευμα η συζήτηση για τι περιοπτώσει παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων να μπει τελευταίο σημείο στην ημερήσια διάταξη και ο κύριο Πρέντα θα πάρει το λόγο για να λογίσει το αίτημα. Έχετε το λόγο, κύριε Πρέντα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν είναι η πρώτη φορά που θέτουμε αυτό το αίτημα, πάντα για τον ίδιο λόγο. Παραδοσιακά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τοποθετεί το, την πέμπτο απόγευμα για αυτά τα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μετακινήθηκε η συζήτηση αυτή για λόγους που δεν καταλαβαίνουμε πολύ καλά στο πρωί της Πέμπτης. Και πρόσφατα ε, προσθέθηκαν άλλες συζητήσεις το απόγευμα της Πέμπτης ε, αντί αυτής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οπότε ζητούμε πολύ απλά να επιστρέψουμε σε, στην παράδοση την οποία ακολουθούσαμε επί πολύ καιρό. Σα ευχαριστώ. Θα ήθελα καλύτερα να πάρει το λόγο υπέρ του αιτήματο Πρέντα. Κατά, παρακαλώ. Ας ψηφίσουμε λοιπόν. Ποιο είναι υπέρ του αιτήματο Πρέντα. Μα σηκώσει το χέρι παρακαλώ. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται το αίτημα. Ω, ήταν σαφές. Εντάξει, εντάξει. Εφόσον ζητείτε έλεγχο, ας κάνουμε εικονικό έλεγχο. Abstimmung ist geschlossen. υπέρ, 205 κατά. Ε, δεν ήταν και ωριακό το αποτέλεσμα. Και έτσι λοιπόν ε, ορίζεται το σχέδιο εργασίας για την τρέχουσα εβδομάδα. Να περάσουμε τώρα στην δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε ό,τι αφορά τη συνάντηση υψηλού επίπεδου του ΟΗΕ για το HIV AIDS. Ο Επίτροπος Άντριο Κάτης έχει το λόγο.